Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασή συνεδρίασής αν συμφωνείτε. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 μας κοινοποιήθηκε με κάποια καθυστέρηση, αντίθετα με την συνήθι πρακτική, βάσει της οποίας το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει το σχέδιο ε, στα μέσα Μαΐου για να επιληφθεί απευθείας και το κοινοβούλιο του σχεδίου. Χαιρετίζουμε τον γενικό μας ε, εισηγητή. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Υπενθυμίζω, όπως έλεγα, ότι ήταν μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε για την κοινοποίηση του σχεδίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπρεπε κανονικά μας κοινοποιηθεί πριν την 30 Ιουνίου και κατά πάσα πιθανότητα γι' αυτό είχε οριστεί και το δημοψήφισμα για το Brexit 23 Ιουνίου. Συμφωνήσαμε λοιπόν εκτάκτως να οργανώσουμε αυτή την σύσκεψη διότι η κυρία Γεωργίευα ήταν πολύ σύντομη στην παρουσίαση του σχεδίου και χρειαζόμασταν κάποιες μέρες για να ανταλλάξουμε ιδέες για το σχέδιο προϋπολογισμού. Εάν δεν έχετε παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσια διάταξης και στο πλαίσια των ανακοινώσεων του Προέδρου σας ε, ενημερώνω ότι αποφάσισαν οι συντονιστές να ζητήσουν βάση του άρθρου 54 και επί της πρωτοβουλίας ε, της Επιτροπής ε, ΡΕΤΖΙ σύνδεση με την Επιτροπή για τα νέα μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Θα περάσουμε τώρα στο σχέδιο προπολογισμού για το 2017. Ο Γιάννης Κάιερ έχει το λόγο με την ιδιότητα του Γενικού Εισηγητή θα κάνει μια γενική αποτίμηση του σχεδίου προϋπολογισμού. Φυσικά είναι ιδιαίτερα αισθητή η μείωση των πιστώσεων πληρωμών προς μεγάλη μας έκπληξη. Διαπιστώσαμε επίση ότι κινητοποιείται ένα, ε, ένα αποθεματικό για τη γεωργία και για την διοίκηση αρκετά μεγάλο. Ε, Γενική Συγητή, έχετε το, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καθυστέρησα επειδή κάθισα και κοιτούσα τις ε, σημειώσεις μου. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι σήμερα το βράδυ δεν θα μπορέσω να σας δώσω την πλήρη επισκόπηση γιατί το πράγμα είναι λίγο περίπλοκο, υπερβολικά περίπλοκο. Αλλά να κάνουμε κάποιες Πρώτες παρατηρήσει. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και κάποια ζητήματα τα οποία καλό θα κάνουμε να τα συζητήσουμε, όπου και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις ε, των άλλων ε, σκιωτών εισηγητών των άλλων ομάδων, γιατί θα πρέπει από κοινού να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική ε, του Κοινοβουλίου. Ένα, Α, δύο και 4. Αυτές τις, αυτούς τους τομείς κοίταξα καταρχάς στο 1α. Ήδη στην πρόταση του προπολογισμού του είδαμε ότι είναι πολύ περιορισμένο το α, περιθώριο, 81 εκατομμύρια και το μεγαλύτερο τμήμα των πληθυκών προγραμμάτων και των προγραμμάτων αυτών θα χρηματοδοτούνται. Το θέμα λοιπόν που πρέπει να απαντήσουμε το είπα και την προηγούμενη Πέμπτη, είναι κατά πόσον θέλουμε να αφήσουμε αυτή την διακοσμητική, αν θέλετε, φύση σε περιθώριο ή αν θα θέλουμε να εξαντλήσουμε το ανατόριο του δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω δεν είναι άποψη της ομάδας μου αυτό, αλλά είναι δική μου προσωπική άποψη και ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι είμαι κάπως επιφυλακτικό σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης να καταστεί αυτό η νέα μηχανή της ενσωμάτωση τη ενοποίηση. Αυτό όμω είναι γενικής φύσεως πολιτική παρατήρηση. Και τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο να... σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ε, τέτοιων μέτρων και για την άμυνα ε, όταν ήδη είναι υπερβαρημένος ο προπολογισμό. Και στην αποσύνδεση των ε, ε, project της ΚΕΠΑ θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτά τα πολύ ακριβά ποιοτικά προγράμματα θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε από τις ίδιε πηγέ όπως και τα άλλα προγράμματα και έχω και θέματα επί της αρχής σε ό,τι αφορά την προσέγγιση όπω σα είπα. Είμαι ικανοποιημένο που στο 1α έχουμε ε, ίδιες υποχρεώσεις και ε, δεσμεύσεις 10,9 και 11 εκατομμύρια. Θα πρέπει να δούμε πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δαπανίσει τα χρήματα αυτά και κατά πόσον θα ανταποκρίνεται στις δικές μας προτεραιότητες. Αυτό που είναι σημαντικό στην ε, φάση αυτή είναι να μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν με τον προπολογισμό αυτό, όπως έχει συμφωνηθεί, να διαθέσουμε τα 2,641 ε, ε, δισεκατομμύρια εγγύηση και 2,3 δισεκατομμύρια πληρωμές. Αυτά λοιπόν θα προέλθουν από τα μη εξαντλημένα περιθώρια και 85 από το Ράζονινγκ 2020 και 120 από άλλα προγράμματα. Είναι σαφής λοιπόν η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ασκήσαμε κριτική και θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε σε αυτή τη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού τι μπορούμε να κάνουμε το Connective ε, Europe Facility και το Horizon 2020, ε, πώς μπορούμε να μην τα εξαντλήσουμε αυτά. Το τόνισα αυτό και στην Ολομέλεια, αλλά θα ήθελα να ακούσω και ποια είναι η άποψη των ε, άλλων ομάδων ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευράς μας από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ε, μας ε, ασκείται και κριτική σε ό,τι αφορά την απόδοση του ΕΦΣΥ. Όχι τόσο το γεγονός ότι υφίσταται και υπάρχει. Αυτό είναι βούληση του Κοινοβουλίου και της ομάδας μου, αν μου επιτρέπετε να τονίσω ούτε απαραίτητα το πώς χρηματοδοτήθηκε, αλλά το performance, η απόδοση, η αποδοτικότητα του ΕΦΣΙ. Αυτή μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω, γιατί τίθεται το θέμα της συμπληρωματικότητα, το οποίο στην παρούσα φάση δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό, σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και λοιπόν ανακύπτει το ερώτημα το κατά πόσον η ΕΤΕΠ με τα χρήματα αυτά και σε ό,τι αφορά τι εγγυήσει των πιστώσεων που δίνει, μήπω κάνει τελικά αυτά που έκανε έτσι κι αλλιώ. Έχουμε μια κοινή έκθεση πρωτοβουλία, λοιπόν, που θα κληθεί να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Και θεωρώ ότι η έκθεση πρωτοβουλία αυτή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα. Να περιμένουμε λοιπόν πρώτα την έκθεση πρωτοβουλία και μετά να κάνουμε σχόλια και παρατηρήσεις προς την Κομισιόν και προς την ΕΤΕΠ. Η ΕΤΕΠ θα παρουσιάσει μια έκθεση για, για το ΕΦΣΙ αυτή την εβδομάδα και θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν και εμείς πώς τοποθετείται και τι επιχειρήματα χρησιμοποιεί και η ίδια η ΕΤΕΠ για το θέμα της συμπληρωματικότητας. Δεν πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν κοιτεθεί για το ΕΦΣΙ θα πρέπει να διαγραφούν από τον προπολογισμό, αλλά δύο φορές ήδη έχω πει ότι μπορούμε και πρέπει να σκεφτούμε το κατά πόσον οι πόροι αυτοί θα πρέπει να μπουν σε ένα μεγάλο βαθμό στο παθηματικό. Μέχρι να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις από την ΕΤΕΠ και από την Κομισιόν και να πιστούμε για την συμπληρωματικότητα και τα κίνητρα. Στη, στο 2 τώρα. Στο τίτλο 2 λοιπόν. 5,7% μείωση συνολικά περιθώριο 1,3 δις περίπου. 650 εκατομμύρια για το contingency margin και για την ενίσχυση του τίτλου 4. Δεν θεωρώ ότι είναι δραματική αυτή η περικοπή, γιατί έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις του 2014 που αναπρογραμματίστηκαν για την ανάπτυξη της υπέτρα του 2016. Αυτό θεωρώ ότι γενικά θα δώσει ε, μια ανακούφιση ε, στην αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε μια πόλια 1,1 δις ε, σε ό,τι αφορά τον γαλακτοκομικό κλάδο και τα έσοδα αυτά. Και πολλοί που είναι στην Επιτροπή Γεωργίας πιστεύουν ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν στον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης και ότι ο κλάδος χρειάζεται κατεπίγοντος τα χρήματα αυτά. Ε, Υπάρχουν και φυσικά αποθυματικά στα περιθώρια που προβλέπονται. Σε ό,τι αφορά την αλληλεία τώρα, θα ήθελα να κοιτάξω την χρηματοδότηση. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν αρκετά χρήματα για τις ειδικέ σχέσει για την βιωσιμή αλληλεία. Αυτό που λέμε εμείς ε, συνέχεια και επανειλημμένα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει και να καταπολεμήσει τις ε, αιτίες ε, των προβλημάτων και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και την βιώσιμη αλληλεία και τις ε, τοπικές ε, ενώσεις ε, αλληλείας. Το θέμα είναι κατά πόσον η μεταρρύθμιση στον τομέα της αλληλείας που έγιναν από νομική άποψη μπορούν να λειτουργήσουν και από χρηματοδοτική άποψη. Γιατί μόνο μία νομική διάταξη, η οποία σε τελική ανάλυση ε, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα, αυτό δεν είναι καλό φυσικά ούτε για τους ελείς, ούτε και για τα ψάρια. Αν θέλουμε λοιπόν να σταθεί με επιτυχία η λευτική πολιτική, θα πρέπει να φροντίσουμε τα εργαλεία της κοινή ελευτική πολιτικής να λειτουργούν για το life. Ε, τα έξοδα είναι πιο υψηλά από το 2016, καλό αυτό. Μας ικανοποιεί να δούμε και τι έγινε. Θα κάνει και το Συμβούλιο, γιατί την τελευταία φορά Έκανα και περικοπέ. Τώρα, στον τίτλο 4, το πιο σημαντικό σημείο το οποίο θέλω να συζητήσω μαζί σα σε παρόμοια η κατάσταση, όπω και στη Γεωργία, σε ό,τι αφορά τι πληρωμέ. Έχουμε ποσοστιαία μείωση, αλλά οφείλεται στο γεγονός αυτό ότι στο παρελθόν είχαμε τόσο μεγαλύτερη αύξηση. Πέρσι λοιπόν, οι πληρωμές ε, στον τίτλο 4 αυξήθηκαν κατά 36% για λόγους που θυμάστε όλοι καλά. Άρα, σε σχέση με αυτή την ε, πολύ μεγάλη αύξηση πέρσι ποσοστιαία, έχουμε 8,5% μείωση, αλλά και πάλι είμαστε πολύ πιο, σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι παλιά. Λόγω της πολιτικής κατάστασης. Τώρα, κατά πόσον οι πληρωμές μπορούν να αποκριθούν στο επίπεδο αυτό. Ε, αμφιλεγόμενο αυτό σήμερα και υπάρχουν και επιχειρήματα. Γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε από κοινού πώς η υλοποίηση των project των Trust Funds θα αναπτυχθεί το 2016. Αυτό τι σημαίνει, κατά πόσον θα αδειάζουν πιο γρήγορα τα Trust Funds αυτό θα ήταν θετικό υπό την έννοια ότι θα κάναμε κάτι για τους πρόσφυγες και για την καταπολέμηση της, ε, των αιτιών που ο κόσμος φεύγει από τις αιστείες του. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω, θα πρέπει να την ε, δούμε και με λίγο δισταγμό. Ο τίτλος 4 εξαρτάται πάρα πολύ και από την δεύτερη δόση της, ε, των πληρωμών για την ευκόλυνση για την Τουρκία. Ξέρετε ότι τρίτα τέταρτα του ποσού αυτού για το οποίο έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή η Ένωση, 750 εκατομμύρια δηλαδή. Για τα 750 λοιπόν αυτά εκατομμύρια προκειμένου να τα διαθέσει η Κομισιόν έχει περικόψει όλες τι υπόλοιπε δαπάνες για τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία. Άρα τα χρήματα αυτά προέρχονται κυρίως από την προενταξιακή βοήθεια υποχρεώσει σχετικέ αυξάνονται κατά 20% και έτσι 72 εκατομμύρια έρχονται από το DCI, το εργαλείο DCI 3,1% αύξηση το εργαλείο που συνδράμει στην σταθερότητα για... και εδώ λοιπόν και από εδώ α, παίρνουμε 65 εκατομμύρια για την διευκόλυνση για την Τουρκία. Και κάτι το οποίο με δυσαριστεί ιδιαίτερο στο Ευρωπαϊκό Εργαλείο μέσω για την γειτονία παραμένει στο επίπεδο του 2016 και γίνεται μια ιστορική ανακατάρταξη και ε, η γραμμή για τη Μεσόγειο για την πολιτική γειτονία μειώνεται κατά 2,4% και τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε για τον ΟΗΕ για την Παλαιστίνη ε, μειώνεται κατά 2,7%. Από τη διάσκεψη του Λονδίνου από την οποία αποτύχεται θα ωφελούνταν και ο Λίβανος και η Ορδανία που φιλοξενούν πάρα πολλούς πρόσφυγες από τη Συρία. Αυτό λοιπόν είναι λίγο δύσκολο θεωρώ και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζουμε τους πρόσφυγες σε μια χώρα αλλά ε, για αντιστάθμισμα ε, ρίχνουμε εντελώ κάποιες άλλες χώρες οι οποίες επίσης ε, έχουν πολλούς πρόσφυγες και άρα ουσιαστικά αυτό τι κάνει, κινητοποιεί άλλο ένα ρεύμα προσφύγων. σε ό,τι αφορά και τους Παλαιστινίους και το, την Ούνδρα. Διαπιστώνεται ότι όταν ε, ο Ούνδρα του ΟΗΕ δίνει δυνατότητες επιβίωσης και κάποια βασικά χρεώδη στα παιδιά, ο κόσμος μένει στις αιστείες τους. Η ανθρωπιστική βοήθεια μειώνεται κατά 14,7% ε, σε ό,τι αφορά το 2016 όμως υπήρχε μεγάλη αύξηση τα περασμένα έτη και αυτό από, ε, από προπολογισμού δεν αποτελεί πρόβλημα και μπορούμε να ενισχύσουμε το θέμα αυτό της αναπτυξιακής βοήθειας από τον προπολογισμό, από το παθηματικό. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας εργασίας σε ό,τι αφορά τη συνολική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ε, χρηματοδοτούμε ένα ολόκληρο τέτοιο ζήτημα από το παθηματικό. Προσοχή. Αυτή ήταν τρει από του βασικότερου τίτλου που ήθελα να αναφέρω σήμερα το βράδυ. Να ευχαριστήσω και την γραμματεία γιατί μας ε, κάνανε κάποιε παρατηρήσει για το πώ μπορούμε να κινητοποιήσουμε κάποιου πόρου στον τίτλο 4. Αλλά θα ήθελα να το συζητήσω αυτό για την κινητοποίηση των επιπλέον πόρων και μαζί σας. Ευχαριστώ. Merci, monsieur le rapporteur. Σας ευχαριστούμε, Γενική Συγητά, και για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ανάλυση, για, τα υπόλοι... για τους υπόλοιπους τίτλους θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ. Για τα άλλα τμήματα, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουμε εγκρίνει εδώ στην Κοινοβούλια, αυτό που μας αφορά εμάς και συνεχίζονται οι ανταλλαγές με το Προεδρείο βάσει του ιστορικού κανονισμού για όλες τις διατάξεις, σε όλα τα άρθρα. Αργά ή γρήγορα θα μάθουμε ποιοι είναι η έκφραση των συζητήσεων. Ε, οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο και δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Επιτροπή των Περιφερειών μέχρι και ε, δικαστήριο. Έχω έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους και θα πρέπει να αναλύσω την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν σε ε, ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν πως θα πρέπει να περιοριστώ σε αυτά τα λιγοστά σχόλια. Ακόμη και αν υπάρχουν ερωτήσεις, σε 9 στις 10 δεν θα είμαι σε θέση να τις απαντήσω, ας το λέω. Ευχαριστούμε που δεν αφήσατε καμία αμφιβολία ε, θα συναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα με το Γενικό Γραμματέα. Θα απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας, σίγουρα. Καλώ τους κύριους εισηγητές τώρα του προϋπολογισμού για το 2017 να μας παρουσιάσουν την ανάλυση τους. Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής, αλλά θα σας δώσω μια πρώτη έτσι, εικόνα αντικαθιστώντας τον συνάδελφο που ήταν στη συνεδρίαση κανονικά και θα έπρεπε να μιλήσει, αλλά τώρα ε, βρίσκεται στην Ολομέλεια για να εκφράσει εκεί την άποψή του. Μία άποψη η οποία δεν είναι καθόλου αντίθετη με αυτή που θα σας παρουσιάσω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση στις πληρωμές κατά 6,2% στον προϋπολογισμό του 2017. Αυτό σημαίνει ένα απλό πράγμα. Σημαίνει ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι στο ύψος που θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν για να εκτελέσουν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που ξεκινάει το 2014 και πάει μέχρι το 2020. Προσοχή, προσοχή. Το 2017 είναι η τέταρτη χρονιά, αν αρχίσουμε το μέτρημα από το 2014. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα έχουμε τεράστια προβλήματα με τις πληρωμές μετά το 2017. Πρέπει να είμαστε σαφείς και να περάσουμε πάρα αυτό το μήνυμα. Να πούμε δηλαδή ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθυστερεί, θα πρέπει να επιταχύνουμε την εκτέλεσή του και αυτή η μείωση που παρατηρούμε σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, θα την πληρώσουμε ακριβά. Πρέπει να, γίνει μια, να υπάρξει μια αύξηση. Να σας θέσω ένα ερώτημα. Είμαστε σε υστέρηση, σε καθυστέρηση, γιατί υπάρχει διοικητικό πρόβλημα, υπάρχει δυσκολία να δρομολογηθούν τα προγράμματα ή γιατί τα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσδοκούσαν τα κράτη-μέλη ή γιατί σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει πρόβλημα εξασφάλιση χρηματοδότηση. Γιατί η χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, όπω ξέρετε, δεν καλύπτει το 100% των αναγκών. Και ίσω κάποια κράτη-μέλη διστάζουν να δανειστούν. Όχι, δεν οφείλεται στο δανεισμό. Θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονό ότι υπάρχει πρόβλημα και με τους κανονισμούς αλλά και με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει πρόβλημα με τις διαδικασίες. Ε, οι, δια, οι συμφωνίες σχέσης, ας πούμε, είναι πολύ χρονοβόρες. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να μπουν στο αυλάκι. Αλλά κοιτάξτε, η πολιτική συνοχής, Φερρυπίν, θα, θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί θα δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τις πληρωμές. Και μία μείωση των πληρωμών σημαίνει αργότερα μία αναγκαστική αύξηση, πολύ μεγαλύτερη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να παρατηρήσουμε τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Δεύτερον, να είμαστε προορατικοί και να κάνουμε έναν σχεδιασμό ό,τι αφορά τις πληρωμές στο μέλλον, γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι σε λίγο χρόνο θα έχουμε περισσότερες, ε, θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών από τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Θα ξεπεράσει δηλαδή το πρώτο κομμάτι πιστώσεις πληρωμών, θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις υποχρεώσεις. Επίσης, Έχουμε μικρή εκτέλεση των πληρωμών και αυτό σημαίνει ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθυστερεί, καθυστερεί η εκτέλεσή του και η συνέπεια είναι αυτή που σας είπα. Ο προϋπολογισμός του 2017 θα πρέπει να είναι ένας προϋπολογισμός συνεπής ως προς τις θέσεις που έχουν ε, ληφθεί συνενετικά. Ακόμα και για την αθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου υπάρχει συνένεση. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι δεν συμφωνούμε με αυτέ τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει στον προπολογισμό, αφού έχουμε δεσμευτεί ήδη στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν γίνονται αυτά. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε επίση. Αλλά διαφωνώ ω προ το πώ αντιμετώπισε διάφορα πράγματα. Αν αρχίζουμε τις επιμολύσεις του προπολογισμού και βάλουμε διάφορα θέματα εκεί, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύση και δεν θα συζητήσουμε ποτέ τα ουσιαστικά. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικές, Στρατηγικών Επενδύσεων ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε μία θέση, έχει μία θέση το Κοινοβούλιο, και για το ορίζοντα 2020 και για το Connecting Europe Facility, ε, το μηχανισμό διευκόλυνσης της το μηχανισμό ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Επίσης, ε, το θέμα είναι όχι μόνο ο προπολογισμό, είναι το θέμα τη προσθετικότητα. Θα πρέπει να υποχρεώσουμε ο κανονισμό που υιοθετήθηκε να γίνει σεβαστό οι κανονισμοί. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα, έχουμε μία, θα, θα συντάξουμε μία έκθεση μαζί με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, την ΕΚΟΝ και θα κάνουμε τις απαραίτητες αξιολογήσεις. Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε αυτό το ταμείο ω προτεραιότητα στις συζητήσει που θα κάνουμε για τον προπολογισμό, το Ταμείο δηλαδή ε, Στρατηγικών Επενδύσεων. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την εκτέλεση, αλλά μην ξεχνάτε ότι το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο δηλαδή Στρατηγικών Επενδύσεων, μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να κινητοποιήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη ανησυχία των πολιτών είναι φυσικά η απασχόληση και κυρίως η απασχόληση των νέων. Αλλά ανησυχούν επίσης και πώς θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Και γι' αυτό δεν βλέπω μάσχημο μάτι την πρόταση της Κομισιόν για να υπάρξει μια προπαρασκευαστική δράση, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη των πολιτών και να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια. Δεν θέλω να πω σε κάθε τίτλο, αλλά πάντως αυτά που ακούσατε τα είπα έτσι γενικά. Και είμαι πεπισμένος ότι με τον γενικό εισηγητή μας και με τους κοιότης εισηγητές θα κάνουμε μια δουλειά στο ύψος των περιστάσεων. και των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εισαγωγική του αυτή παρατήρηση γιατί νομίζω ότι είμαστε διαφώτισε αρκετά. Εμεί πάντα ξεκινάμε με ένα σχέδιο προϋπολογισμού και προσπαθούμε λοιπόν να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση κατά πόσον μπορούμε να ξεσκονίσουμε διάφορα σημεία. Νομίζω ότι έχουμε πλέον ένα σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο καταρχάς προσανατολίζεται στην πραγματικότητα. Θέτει σωστέ προτεραιότητες και νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να το τονίσουμε αυτό επανειλημμένα. Επιτέλους στον ε, τομέα της μετανάστευσης ξεκινάμε να καταπολεμούμε τα βαθύτερα αίτια και να προβλέπουμε μέσα με τον προπολογισμό γιατί είναι σαφές ε, για όλους μας ότι θα μπορούσαν να είναι και, πολύ, και, και μεγαλύτεροι οι δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη πιστεύω ότι και εδώ, σε αυτόν τον τομέα, πρέπει αναγκαστικά και υποχρεωτικά παράλληλα να έχουμε και ένα συνολικό όραμα προκειμένου στην τελική ανάλυση οι πόροι αυτοί να δαπανηθούν με τον βέλτιστο τέτοιο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει για μένα ε, συγκεκριμένα. Δεν βλέπω να υπάρχει μία συγκεκριμένη ε, κατεύθυνση ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι το νομικό πλαίσιο, ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ, πώ θα ασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι απόλυτα σύμφωνο να δαπανηθούν πιο πολλοί πόροι. Αλλά αν ε, μεταφερθώ στη θέση ενό φτωχού σνοριοφύλακα, αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται απίστευτα να πετύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ω εκ τούτου, πιστεύω ότι πέρα από τα μέτρα, τα μέσα του προπολογισμού, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και η σωστή, να υπάρχει το σωστό νομικό πλαίσιο. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερο και ε, δεδομένου του Brexit, να, θα πρέπει να μην ε, μπει στη γωνία, θα πρέπει επιδετικά να ακολουθήσει μια σωστή πολιτική. Και έτσι μπορούμε να πείσουμε, θεωρώ, και τους νέους και όλους τους πολίτες της Ένωσης ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Σωστό λοιπόν είναι το γεγονός ότι προβλέπονται πόροι από τον προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το σωστό πλαίσιο για να μην ξοδέψουμε ε, χωρίς αποτέλεσμα πολλά χρήματα. Κάτι άλλο. Με παρόμοια επιχειρηματολογία. Θα ήθελα να επαναλάβω την κριτική που έχω ασκήσει επαναλημμένα για το ΕΦΣΥ. Εγώ πιστεύω, αντίθετα με τον συνάδελφο Φερνάντε, ότι ασφαλώς μπορούμε να πούμε ότι 100 δισεκατομμύρια έχουν δαπανηθεί και ότι αυτό είναι σήμα ποιότητας. Αλλά αν θέλουμε συνολικά να προκαλέσουμε επενδύσεις 300 δισεκατομμυρίων, έχουμε φτάσει μόνο στο 1 τρίτο. Και ως Επιτροπή Προπολογισμού θα πρέπει τώρα να ασχοληθούμε πολύ α, με το τι έχουμε πετύχει. Α, και το σκέλος της ε, συμπληρωματικότητας, πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς έγιναν οι επενδύσεις. Ήταν άμεσα, έμεσα από το δημόσιο μήπως τομέα, γιατί αυτό θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι τα κράτη, οι δήμοι που έχουν δαπανίσει έχουν αυξήσει το χρέος τους. Αυτό θέλουμε, να αυξήσει το χρέος, το δημόσιο. Και ιδιαίτερο ό,τι αφορά τι χώρε τη Ευρωζώνη, υπάρχει και του Μάστρετ με συγκεκριμένα κριτήρια, η οποία δεν τηρείται. Τα κριτήρια αυτά δηλαδή. Ε, τέτοια λοιπόν ε, ζητήματα δεν μπορούμε να τα αγνοούμε σε τέτοιε εκθέσεις γιατί είναι και αυτά ένα σημαντικό ζήτημα. Και για λόγους σαφήνειας, θα ήθελα να μην πούν από την πίσω πόρτα με μικροποσά ε, προγράμματα όπως η Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί. ενδεχομένω να καταλήξουμε μετά από συζήτηση, δημόσια συζήτηση, ότι τα χρειαζόμαστε τα προγράμματα αυτά και ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη. Αυτό εντάξει, αλλά όχι από την πίσω πόρτα. Ε, και άλλα πολλά θα είχα να πω, αλλά θα περιοριστώ σε αυτά. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη όλους, από όλους τους κυρίως από το Γενικό Εισηγητή, γιατί ε, ήμουνα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, είχαμε ψηφοφορίες και δεν τον άκουσα. Αυτή είναι και η τιμωρία σας, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω μία σκέψη για τον ΤΑΚ 3, το προσχέδιο προπολογισμού 3 του 2016 που ε, είναι σωματωμένο στο γενικό πίνακα που μας έδωσε η Κομισιόν για το σχέδιο προπολογισμού του 2017. Εκεί δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Βλέπουμε ότι έχουμε, έχουμε λάβει υπόψη τα ε, αιτήματα των διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων για την ασφάλεια. Ε, ήδη στο προϋπολογισμό του 2016 είχαμε προβλέψει 15 εκατομμύρια. Το ερώτημά μου είναι τι γίνεται με τις πιστώσεις, τις έκτακτες πιστώσεις που είχαμε ψηφίσει έχουμε περισσότερες ανάγκες μετά από τις απόπειρες τις τρομοκρατικές. Ε, τι γίνεται με την ε, κατανάλωση, με το ξόδεμα αυτών των ποσών. Ε, γιατί το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Πρόκειται ε, για τη δημιουργία 35 επιπλέον θέσεων για να βρούμε ε, άτομα για την ασφάλεια, ούτως ώστε να έχουμε ένοπλη προστασία σε στρατηγικά σημεία στο εσωτερικό των τριών κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι υπέρ των ενέοπλων αυτών ατόμων. Έχετε πάει σε άλλα τμήματα τώρα του πίνακα, έτσι. Ναι, μιλάω για τα άλλα τμήματα. Αλλά επειδή μιλάμε για τον προπολογισμό του 2016 και εγώ ήμουν εισηγητή για τον προπολογισμό του 2016 και η Κομισιόν έχει βάλει αυτό το σημείο στο γενικό τη κείμενο για τον προπολογισμό του 2017, ε, τι ρωτώ με, πούμε, τι νόημα έχει αυτό. Θέλω να επανέλθω, Πρόεδρε, σε κάτι. Δεν είμαι κατά, αλλά είμαι υπέρ του συστήματος που προβλέπετε. Ούτε, για, ούτε η, γιατί ούτε η βελγική χωροφυλακή, ούτε ε, ο στρατός του Βελγίου μπορούν να μπουν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, αν μπουν τρομοκράτες ε, μέσα στα κτίρια μας, δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Εάν η χωροφυλακή των Βέλγων ε, εμποδίσει όμως τους τρομοκράτες να μπουν στο Κοινοβούλιο, ε, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα. Ναι, αλλά πρώτα δεν μπορεί να συμβεί επίθεση στο Στρασβούργο έτσι, ή στο Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστώ για αυτό το, το σχόλιο το οποίο το, με το οποίο θέλετε να με κολλήσετε στον τοίχο, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Αστιάκι τώρα ήταν αυτό. Τέλο πάντων, είναι ε, ιδιάζων αυτός ο μηχανισμός. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό ε, νομικά στο, στην βελγική επικράτη χωρί συμφωνία με το βελγικό κράτος. Γιατί έχουμε μέσω του συστήματος προνομίων και ασυλίας, α πούμε, διάφορε ε, κάποιε ειδικέ μεταχειρήσει, α πούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Έχουμε ε, συμφωνήσει τίποτα με τι αρχέ των διαφόρων ε, χωρών. Επίση, επί χρόνια τραβούσαμε τα μαλλιά μα για να πετύχουμε αυτή τη μείωση του 5%. Για αυτή τη μείωση του 5%. Τι θα κάνουμε τελικά, θα το βάλουμε στο 5% αυτά τα ποσά, ε, θα τα αφαιρέσουμε, ε, θα έχουμε επιπλέον ε, οδηγού οι οποίοι δεν θα είναι υπάλληλοι όμω. Δηλαδή ή θα είναι ειδικέ θέσει αυτές που δεν μπαίνουν στο, γενικούς, ε, ε, στο γενικό προϋπολογισμό. εδώ όμως μιλάμε για θέσεις RD5, άρα μιλάμε για υπαλλήλου, έτσι. Τώρα, οι επιπλέον πιστώσεις χρειάζονται. Ε, είναι γελίο. 225 εκατομμύρια ευρώ Τα άλλα ε, θεσμικά όργανα ζητάνε τελείω άλλα ποσά. Τι παίζεται εδώ πέρα. Επίσης, τι γίνεται με τις συμφωνίες με τις εθνικές αρχές. Ε, καλύπτονται αυτές οι συμφωνίες από το σύστημα προνομίων και ασυλιών. Και τρίτον, όλα αυτά έχουν να κάνουν τον προπολογισμό του 2017. Τούτου λεχθέντος θέλω να επανέλθω σε ένα σημείο το οποίο έθιξε ο κύριος Φερνάνδης, ο οποίος στο μεταξύ έφυγε δυστυχώς. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο είναι περίεργο σε αυτό που μας προτείνουν ότι αφορά τις πληρωμές. Θα θυμάστε ότι όταν ε, είχαμε την κρίση με τις πληρωμές ε, το 2014-2015, είχαμε πρόβλημα με τον τίτλο 1β. Εκεί είχαμε καθυστερήσει πληρωμών. Κοιτάξτε τον πίνακα. Γιατί βλέπετε. Βλέπετε ότι ο τομέας όπου είχαμε κατάρρευση των πληρωμών είναι 23,5% παραπάνω από ότι όλα τα άλλα ποσά στις άλλους, άλλους τίτλους. επομένως, ή είναι προϋπολογισμός Brexit αυτός, δηλαδή το κάναμε ούτως ώστε να μην ε, τσαντιστούν οι Βρετανοί. Ε, δηλαδή να μην τους ζητήσουμε να περάσουν από το Ταμείο για να ξυλωθούν το 2017 παρότι θα φύγουν ή ξαναδημιουργούμε από την αρχή ε, όλες τις προϋποθέσεις για να προκύψουν αυτά τα προβλήματα που θέλαμε να γλιτώσουμε. Αλλά έχουμε ε, σπείρει του πόρους για αυτά τα προβλήματα ήδη. Τρίτο στοιχείο που θέλω να σας τονίσω είναι ότι καταρχήν συμφωνούμε με τις προτεραιότητες του προγράμματος της Κομισιόν, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καινοτομία και ανάπτυξη. Γι' αυτά μιλάει η Κομισιόν βασικά. Η ομάδα μου δίνει ιδιαίτερη σημασία φυσικά στην εξέταση των προτάσεων υπέρ της καινοτομίας, υπέρ των μικρομέσων επιχειρήσεων και των νέων. Γιατί είναι στρατηγικά στοιχεία, επί των οποίων θα πρέπει να επιμείνουμε. Και το λέω εδώ μπροστά σε όλου του συναδέλφου. Το να πούμε στη, στην κοινή γνώση, γνώμη ότι έχουμε επιπλέον ε, κονδύλια για την μετανάστευση είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν πρόκειται αυτό να συμφιλιώσει τον κόσμο με, την, με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα πρέπει παράλληλα να δείξουμε ότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση δίνει αποτελέσματα. it delivers, όπως λένε οι Βρετανοί, για τους νέους. Και το πρόγραμμα, τα προγράμματα για τους νέους, για μένα, θα πρέπει να είναι ακρογωνίως λήθος των προσπαθειών που θα κάνουμε στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Τώρα για για τη μετανάστευση έχω δεκάδες ερωτήσεις, αλλά δεν θέλω να εκνευρίζω τους συναδέλφους με αυτό το θέμα. Αν εξετάσω προσεκτικά όμως τα σημεία, υπάρχουν θεματάκια που ε, χρήζουν απαντήσεων. Θέλω να μιλήσω για, την, για το EU Λίζα. Ε, είναι το, ο μηχανισμός είναι το 2016 είχε 82 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Για το 2017 153 εκατομμύρια. Μιλάμε για μια αύξηση 91,6%. Αυτός ο οργανισμός διαχειρίζεται την πληροφορική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Υπάρχουν τα συστήματα προ, ε, εισόδου, εξόδου ατόμων κτλ. Αλλά να αυξήσουμε τον προπολογισμό 91,3% πρέπει να κάνουμε κάποιε ερωτήσει. Τι, τι παίζεται. Και είναι μία από τι δεκάδε ερωτήσει που έχουμε να κάνουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά με τη Γενική Γραμματεία για το πώ διαχειρίζεται κάποιε πιστώσει που έχει στη διάθεση το Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη. Ε, εκεί παίζεται ο, το amending budget ε, υπαριθμών 3. Ε, εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εκνοβουλευτικής θητείας, αν συνεχίσουμε έτσι, θα μας γυρίσουν μπούμεραν. Ε, για τις προτεραιότητες νομίζω θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην, στον τίτλο 1α. Και ενώπιον του κόσμου εκεί θα δείξουμε ότι οικοδομούμε το μέλλον των Ευρωπαίων και ότι βοηθάμε τους Ευρωπαίους με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ζητώ συγγνώμη ε, που, έφτασα, που έφτασα καθυστερημένος και θα αναγκαστώ όχι μόνο να... Όχι μόνο έφτασα καθυστερημένος, αλλά θα φύγω και νωρίτερα. Καταλάβατε ότι αυτό μας συναχωρεί απίστευτα, κύριε Ντεπχέ. Συμπάσχουμε. Για τις ε, πιστώσεις πληρωμών θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εκκοινοποιήσει ε, το ε, ποσό των ανεξόφλητων λογαριασμών. Θα πρέπει να έχουμε μία ένδειξη. Τι ακριβώς έχει μείνει απλήρωτο. Δεν είναι δεν μπόρεσε να έρθει. Δεν βλέπω κανέναν από την ε, ομάδα. Ερνέστο Μαραγκάλ. Ευχαριστώ. Στο προπολογισμό έχω την αίσθηση ότι είναι τμήμα του γύρου της Γαλλίας. Είναι ενδιαφέρον ο προπολογισμό, αλλά έχει πολλού αγνώστου παράγοντε. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Συμβουλίου. Από πού θα περάσουμε στο βουνό, δηλαδή με τα ποδήλατα. Και όταν ξέρουμε διάφορα πράγματα, ε, θα πρέπει να δούμε μήπω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κινούνται προ εντελώ αντίθετε κατευθύνσει και θα πρέπει να μετρήσουμε και την απόσταση ανάμεσα σε εμά του δύο. Επίση, λείπουν δύο βασικέ κι άγνωστη Είναι κρυμμένη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την αναθεώρηση του πολιετού ε, δημοσιονομικού πλαισίου και δεν ξέρουμε και τι επίπτωση θα έχει το Brexit. Ακόμα. Μόλι συνέβη εξάλλου. Τουλάχιστον ακόμα δεν ξέρουμε τι συνέπειε θα έχει. Αλλά είναι ανησυχητικό που ήδη από τώρα βλέπουμε πώς με την πρόταση αυτή για τον προπολογισμό αυξάνεται η απόσταση ανάμεσα σε εμά και στο Συμβούλιο. Ε, θα το ψηφίσουμε εξάλλου ως ούπο στην Ολομέλεια. Και αυτή η απόσταση ανάμεσα στους δύο ε, προκύπτει ε, μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν. Αυτός ο προϋπολογισμός επίσης μας δείχνει τη δυνατότητα αξιέπαινη κατά τα άλλα της Κομισιόν για αυτή την προσπάθεια εξισορρόπησης. Ευελιξία, ανάμεσα στην ευελιξία, τα περιθώρια, ε, τεχνικές προσαρμογές, περιθώρια και τα πρόβλεπτα και όλα τα κάνει αυτά για να μην ξεφύγουμε από το πλαίσιο, το ισχύον, ας πούμε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προσπαθεί να μην πάμε σε αντίθετη ε, πορεία σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εντάξει, μπράβο αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό που θα ελπίζαμε. Δηλαδή, βασικά τι περιμέναμε από έναν τέτοιο προπολογισμό. Περιμέναμε να μας δείξει ε, να απεικονίζει, εν μια ευρωπαϊκή αντίδραση στις κρίσεις που ζει η Ευρώπη. Για τις πιστώσεις πληρωμών. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριο Ντεπρέ, πολύ σωστά. Αυτό ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι η έκφραση του πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει προστιθέμενη. Προς, δεν έχει κανένα προστιθέμενο ρόλο, καμία προστιθέμενη αξία. Δεν παίζει το ρόλο που τη αντιστοιχεί. ακόμα και όταν πληρώνει, δεν ε, δημιουργεί τις θέσεις απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη που θα έπρεπε να δημιουργήσει κτλ. Ε, τώρα, κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Κλιματική αλλαγή. Η, Γεωργίευα, η κυρία Γεωργίευα μας είπε ότι το σχέδιο προπολογισμού του 2017 είχε το 20,5% των ε, δαπανών, ε, συμπεριλάμβανε το 20,5% των δαπανών για την κλιματική αλλαγή. Αυτό δεν είναι παρκές. Στην πραγματικότητα έχουμε από τα προηγούμενα έτη συσσωρεύσει καθυστέρηση. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Επίσης είναι σε αντίθεση με αυτά που είπε η Γενική Διεύθυνση Κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να πάμε πολύ πιο πέρα από το 20,5%. Και επίσης είναι αντίθετο σε σχέση με αυτό που είπαν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά στο COP21 στο Παρίσι. Ξεχνάμε όλε τι δεσμεύσει που λάβαμε για τη συνολική περίοδο 2014-2020. Για το ΕΦΣΥ. Συμφωνώ. Ποσοτικά ε, υπάρχει, το φαινόμενο δράγη. Ε, υπάρχουν πολλά λεφτά Είμαστε ικανοποιημένοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ε, προσθετικότητα. Να εξασφαλίσουμε ε, επενδύσεις για έργα πιο επικίνδυνα. Επίσης, κάτι που με ανησυχεί. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να δούμε το κατά πόσον εφαρμόζεται το κριτήριο της προσθετικότητας. Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι θέμα δημοσιονομικό προσθετικότητα και κίνδυνος. Αυτά είναι βασικά κριτήρια και θα πρέπει να τα ε, σεβαστούμε. Εράσμος Erasmus Plus. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και ελπίζω η Επιτροπή Πολιτισμού να μπορέσει να συζητήσει όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και τον προσανατολισμό των αλλαγών και, τον, ε, και τις καθώς και τα, τους στόχους. απασχόληση, νεότητα. Επίσης, εδώ είχαμε κάνει σχετική ε, έκθεση για την ε, αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Το σημείο αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τόσα λέγαμε εμείς σε εκείνη την έκθεση. Άμυνα, ασφάλεια κτλ. κτλ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά από αυτά που μας είπε η κυρία Γεωργίευα τις προάλλες, έλεγε ε, ότι μειώνονται οι υποχρεωτικές δαπάνες για το ίτερ, που την καταλαβαίνουμε. Ε, θα υπάρξει μια ε, μετακίνηση κονδυλίων για προγράμματα υπέρ της άμυνας. Προσοχή, προσοχή. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε διάφορα ερευνητικά έργα για την, ερευνητικά προγράμματα συγγνώμη, για την ενεργειακή μετάβαση. Πρέπει να σταματήσω. Τελειώνω, τελειώνω, πρόεδρε. Για την άμυνα. Πρέπει να βοηθήσουμε και να παίξουμε συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη. Να υπάρξει μια ενοποίηση των προσπαθειών επίσης. Το πρόγραμμα για τη συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, υπάρχει μείωση. Δεν είναι καλά αυτά τα νέα. Και η μόνη αντιστάθμιση είναι η αύξηση των κονδυλίων ε, των προενταξιακών των προεταξιακών συγγνωμικών κονδυλίων. Είναι υποχρεωτική αυτή η εν μέρη αύξηση. Αλλά προσοχή, προσοχή. Στην πραγματικότητα είναι μια αύξηση ε, που δεν εκφράζει πραγματική βούληση για περισσότερη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα για τα οποία θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά θα σταματήσω εδώ. Nous revenir. Ναι, ναι, ναι, κύριε Μαρεγκάλ, θα μα δοθεί ευκαιρία και θα επανέλθουμε. Τζάνι. Ε, Πολύ σύντομα, γιατί οι συνάδελφοι ε, έβαλαν τα, το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Σε όλα τα προβληματικά σημεία στάθηκαν. Ε, σε όλα τα σημεία που θα συζητήσουμε πιο ενδελεχώς, αναφέρθηκαν. Δύο σημεία λοιπόν για μένα. Για τις πληρωμές μίλησε ο κ. Φερνάντες προηγουμένως, αλλά μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι. Για το θέμα των πληρωμών, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω την ψαλίδα που μεγαλώνει ανάμεσα στις ε, πιστώσεις πληρωμών και στις ανάληψεις υποχρεώσεων. Δεν καταλαβαίνω. Ακόμα μία φορά μεγαλώνει αυτή η ψαλίδα. Και πώς έχει, έχει νόημα με αυτή τη στρατηγική μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα των πληρωμών. Ο, ο το έλεγε και θα το πει μάλλον και το είπε μάλλον και η Γεωργίωβα. Ίσως οφείλεται στο ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα, δεν χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα, επομένως ε, μειώνονται οι πληρωμές. Αν όμως τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρήμα, αυτά τα ποσά, το να αυξήσουμε τις ε, πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων δεν είναι ίσω η σωστή στρατηγική. Θα πρέπει να ξαναδούμε τις διαδικασίες χρησιμοποίησης αυτών των κονδυλίων και να αυξήσουμε και το να αυξήσουμε αυτό το χάσμα, αυτή την ψαλίδα, δεν μα βοηθάει. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συμφωνώ με την ανάλυση του, στρατη, του εισηγητή. Με βάση τα στοιχεία που έχει η Τράπεζα Επενδύσεων, ε, είναι σαφές ότι για όλα τα έργα που χρηματοδοτούμε σήμερα ίσως υπάρχει ένα το οποίο μοιάζει να είναι κλασικό, ας πούμε, ότι, ό,τι κάνει ακριβώς και η ΜΠΕΙ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επομένως, το, το στοιχείο της προσθετικότητας δεν το εξασφαλίζουμε έτσι. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε μήπως θα πρέπει να υπάρξει ένα πάγωμα ή να βάλουμε σε αποθεματικό αυτά τα κονδύλια. Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα ποσά ή να αφαιρούμε τέλο πάντων λεφτά από άλλου τίτλου προπολογισμού, όπω έγινε για να χρηματοδοτήσουμε το ΕΦΣΥ, χωρί να έχουμε καμία προστιθέμενη αξία. Τελευταία σκέψη. Είναι οι προσπάθειες που θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεδομένων των χαλεπών καιρών, ίσως καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε σε λίγους τίτλους που μπορούν να μας εξασφαλίσουν αυτή την προσθέμενη αξία. Σήμερα, οι στόχοι που ανέφερε η Κομισιόν είναι ξεκάθαροι και τους συμμεριζόμαστε για αυτόν τον προϋπολογισμό. Το να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες και στις πιστώσεις πληρωμών αλλά και στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στην, ε, στον τίτλο 1α, ίσως αυτό να είναι η νικηφόρα στρατηγική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και το μήνυμα στους πολίτες ότι να, θα κάνουμε τις επενδύσεις που θέλουν. Θα κάνουμε τις επενδύσεις για να υπάρξουν και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Επομένως, νομίζω ότι είναι μια στρατηγική που μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Νομίζω έφυγε. Εξακολουθούμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2017. Οι συντονιστές ακόμη δεν τους ακούσαμε. Thank you very much, and thank... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και έπρεπε να πάω στην Ολομέλεια και ευχαριστώ που δώσατε το λόγο στο Ζωζέ Μανώλη Φερνάντες για, για να τοποθετηθεί. Λοιπόν, λαμβάνουμε γνώση τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εργαλείο για την κινητικότητα και το ε, εφεδρικό ε, περιθώριο ενοχής που έχουμε δείχνει ότι στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου υπάρχει αυτή η επιθυμητή ευελιξία. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε με πόσο μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όλες τις προκλήσεις οποίες πρέπει να αντιπεξέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την αναθεώρηση του πολιετούς θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα για τον προκλεισμό το 2017, ναι, είναι πολύ μεγάλη η κρίση, η προσφυγική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα για την οικονομία και την ανεργία. Γι' αυτό και τίτλοι 1α και 1β ε, είναι το μίσο που πρέπει να δράσουμε για να τονώσουμε την έρευνα, την καινοτομία, την ε, απασχόληση. Χρειαζόμαστε επαρκή κονδύλια στους τίτλους 1α και 1β, κυρίως το 1β ή τα επιχειρησιακά προγράμματα του χρόνου ε, θα λειτουργούν θα τρέχουν πλήρω. Ε, το 23% όμω η μείωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 1Β για το 2017 με ανησυχεί. Ε, και από ό,τι κατάλαβα δεν θα υπάρχουν ε, πλέον απαιτήσει πληρωμών για την προηγούμενη περίοδο 2007-2013, όμω ξανά θα τρέχουν όλα τα προγράμματα πλήρω του χρόνου και με ανησυχεί αυτό. Συζητήσεις που κάναμε το Σεπτέμβρη για τους αναξεόφλητους λογαριασμούς ε, και που θα κάνουμε και φέτος το Σεπτέμβριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήματα και με την αναθεώρηση του πολιετού ελπίζω να υπάρχουν νέες προτάσεις για τη συνέχιση του προγράμματος εγγύηση για την νεολαία και για τις επιστώσεις ανάλυσης υποχρεώσεων για την επόμενη χρονιά. Για τον τίτλο 1α με τον ορίζοντα 2020 βλέπουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας των προγραμμάτων μειώνεται από το 20% που ήταν στην προηγούμενη περίοδο και αγγίζει σχεδόν το 13%. Θα μας λείπουν κονδύλια σε αυτό το τομέα. Μόνο 13% των προγραμμάτων μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε σχέση με το 20% των προηγούμενων ετών καλά προγράμματα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις περικοπές από τον ορίζοντα 2020 για το ΣΕΦ ε, και να εκπληρώσουμε τη δέσμευση που αναλάβαμε σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων του ΕΦΣΥ. Ε, για την υποστήριξη των μικρομεσαίων. Καλωσορίζουμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω μα είπε την περασμένη εβδομάδα, αυτέ είναι που δημιουργούν θέσει αποσχόληση για την οικονομία και γι' αυτό πληρώ, ε, υποστηρίζουμε για το κόσμο την αύξηση των πιστώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων. Ε, μα ικανοποιεί πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία. Τώρα για το εφεδρικό περιθώριο, ξαναλέω, υπάρχουν λιγότερα χρήματα ε, στο εφεδρικό τομείο σε περίπτωση επιδείνωσης ε, της τωρινής ε, κρίσης στη γεωργία που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Ξέρουμε ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και για, την, ε, για το τίτλο 3 ή προς τα πάνω αναθεώρηση των ορίων μάλλον δεν θα καταστεί δυνατή. Αυτό όμως προσμένουμε για τον ε, τίτλο 3 και φυσικά για το Ταμείο για την Τουρκία. Βλέπουμε ότι θα βρεθούν τα κονδύλια. Στη συνέχεια για την ανθρωπιστική κρίση αφενός και αφετέρου υποστήριξη προς τη Νότια Μεσόγειο, όλα αυτά αντιβαίνουν σε αυτά που ανέκαθεν λέγαμε ότι η κατάσταση στις χώρες προέλευσης των προσφύγων πρέπει να ε, βελτιωθεί για να σταματήσουν ε, να αναχαιτιστούν αυτές οι προσφυγικές ε, ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέρσι είδαμε και με το Συμβούλιο ότι η περικοπή των κονδυλίων σε αυτό το τομέα είχαν αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ε, στη Νότια Μεσόγειο πρέπει να υποστηρίξουμε την κατάσταση επιτόπου στις χώρες προέλευση των προσφύγων. Στην Ανατολική Γειτονιά έχουμε την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Αυτέ οι τρει χώρε έχουν υπογράψει σύμφωνια σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, καταβάλουν πολλές προσπάθειες, κάνουν θυσίες οι άνθρωποι για να συσφίξουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ανατολική γειτονία όμως δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες, είναι και η Μέση Ανατολή. Αυτές οι τρεις χώρες ε, πολιτικώς πώς έχουν αποφασίσει να συσφίξουν τους πολιτικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Ανατολική γειτονία. Θα σταματήσω εδώ. Προσβλέπουμε ενυπομονησία στις ε, συζητήσεις ε, των επόμενων εβδομάδων ε, με τους αδέλφους στην Επιτροπή, στις Επιτροπές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πάρα πολλά ήδη. Ε, μπήκαμε σε πολλές λεπτομέρειες των προτάσεων. Εάν θέλω να συνοψίσω με μία φράση αυτόν τον προϋπολογισμό, θα, θα έλεγα ότι είναι στον αέρα είναι σαν να μην μπορούμε να αντιδράσουμε, σαν να μην υπάρχει ευελιξία, σαν να μην έχουμε κανένα περιθώριο. Ε, είμαστε εντελώ ε, ασφικτιούμε, ε, σαν να πνιγόμαστε. Ε, κάπως θα πρέπει να αντιδράσουμε. Το 2017 ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι business as usual. Ε, συνεχίζουμε να κάνουμε τις πολιτικές που κάναμε εδώ και 15 χρόνια, τις οποίες πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως. Φυσικά τη γεωργία πρέπει να τη συνεχίσουμε. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πολιτικές συνοχής, αλλά από το 2008 έχουμε και μια οικονομική κρίση που δεν έχει λυθεί. Και έχουμε και μια προσφυγική κρίση που λίγο την περιορίσαμε, λίγα πράγματα μπορέσαμε να κάνουμε. Έχουμε επίσης και τις τρομοκρατικές ε, επιθέσεις που δεν ξέρω πώς ε, με αυτόν τον προϋπολογισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό που που έκανε η Κομισιόν με τα ελάχιστα λεφτά που στη διάθεσή τη έκανε ό,τι μπορούσε. Ε, δηλαδή τι κάνει, ουσιαστικά μεταφέρει, βγάζει από την αριστερή τσέπη και βάζει δεξιά, α πούμε. Μεταφέρει από εδώ εκεί. Τι να κάνει. Νομίζω ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας ε, ενδιάμεσο προϋπολογισμός. Έπρεπε να τον ε, παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει ήδη να αρχίσουμε από τώρα να συζητάμε την τροποποίηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί αν αρχίσουμε να μεταφέρουμε την ε, αριστερή τσέπη στη δεξιά, να βάζουμε δηλαδή ε, να βάζουμε λεφτά για τους πρόσφυγες και τα βγάζουμε από την πολιτική ας πούμε συνεργασίας, στην πραγματικότητα τι κάνουμε. Ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, να βουλώσουμε τρύπε, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που έχει εμφανιστεί σήμερα, βγάζοντα λεφτά από μια άλλη πολιτική που θα, θα τα στερηθούμε, πούμε, και θα εμφανιστεί ένα πρόβλημα αύριο. με τα εργαλεία που έχουμε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα πρέπει, αυτό που να, πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά είναι να πιέσουμε πολύ το Συμβούλιο. Γιατί με αυτό τον προπολογισμό μας αφήνει στον αέρα πραγματικά, μας αφήνει μετέωρους. Δεν είμαι αισιόδοξη. Και μετά αυτό το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι πεντακάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν ανασκουμποθούμε, δεν πρόκειται να φύγει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Πρωτού εξετάσουμε τα υπόλοιπα τμήματα, θα συνεχίσουμε με τον προϋπολογισμό του 2017. Α, και η κυρία Τόμα. Κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Πρωτού ε, μπούμε σε άλλε λεπτομέρειε, να πω δύο λόγια για αυτά που είπε ο κ. Γκάιερ. Θυμόμαστε ότι πριν από κανένα δύο εβδομάδε ε, ψηφίστηκαν κάποιε μεταφορέ, ε, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μειώθηκαν ο αριθμό των διερμηνέων και τώρα βλέπουμε ότι αυξάνεται πάλι ο αριθμό των δερμηνέων και των μεταφραστών. Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι πολύ σοβαρό και αξιόπιστο. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς ε, λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν αυτά τα πράγματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί στη τελική ανάλυση μιλάμε και για την αξιοπιστία μα Τώρα για το γενικό προπολογισμό, Όπω τον πρότεινε ο κύριο Γκάιερ. σε κάποιες ε, περιπτώσεις νιώθω ότι δεν έχουμε άλλο αέρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεργία, ύφεση, τελμάτωση, ιδιαίτερα όλα αυτά πλήττουν τους νέους και χρειαζόμαστε λοιπόν οικονομική αναπτύξη. Γι' αυτό λοιπόν κάτι θα πρέπει να κάνουμε, κάτι πιο αποτελεσματικό, μια πιο αποδοτική πολιτική συνοχή, πιο πολύ προστιθέμενη αξία. Αλλά πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά, καθυστερήσεις, ε, με όλα όσα κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε ανάληψη υποχρεώσεων, ακούσαμε, αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται καλές υποχρεώσεις για να μπορούν να υλοποιούνται καλά προγράμματα. Αν δεν υπάρχουν καλές ε, δεσμεύσεις και ανάληψη τέτοιων ε, δεσμεύσεων, θα παραμείνουν πόροι, οι οποίοι δεν θα αξιοποιούνται. Και αυτό φυσικά θα είναι ει βάρο της υλοποίησης, ει βάρο της εφαρμογής. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πιο πολλέ επενδύσει. και αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε με μια καλύτερη πολιτική συνοχή, αλλά προ αυτή την κατεύθυνση έχουμε και το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Με το Ταμείο αυτό λοιπόν υλοποιούνται τέτοιε επενδύσει. Τέτοιε επενδύσεις όμω που θα υλοποιούνται ενδεχομένω και χωρί το Ταμείο αυτό. χρηματοδοτούνται για παράδειγμα σε κάποιες χώρες κάποια οικολογικά προγράμματα. Πολύ καλά τα λέω, αλλά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και χωρίς το, το ΕΦΣΥ. Χρειάζεται λοιπόν μια ανάλυση του τι χρηματοδοτεί και τι θα έπρεπε να χρηματοδοτεί το ΕΦΣΥ για να μην αφαιρούνται τελικά πόροι από τον ορίζοντα 2020, από το Connect Europe Facility και το καθεξής. Κάτι άλλο που χρειαζόμαστε. Ε, έγκυρες Γιατί αναφέρθηκε ότι όταν το 2017 έχουμε χαμηλές ε, πληρωμές, θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και το 2014 και έτσι θα μείνουν πολύ ανοιχτοί λογαριασμοί και σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα είχε αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές. Σε ό,τι αφορά την ε, ψήφιση τη συντολή των τριμερών διάλογων, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία ανάλυση για τις καθυστερημένες πληρωμέ. Και ως τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα από αυτά που έχουμε ζητήσει. Αν δεν πληρώνονται λογαριασμοί, οι πιστωτές αναγκαστικά ενδεχομένω θα έχουν και αυτοί προβλήματα με την πληρωμή των λογικών τους λογαριασμών, θα απολύουν προσωπικό. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο δύο χρόνια αργότερα καλούμαστε πάλι να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια σωστή ανάλυση της πολιτικής που χρειαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Κεντρική Τράπεζα μας βοηθούν με χαμηλά επιτόκια. Χορηγούν χρήμα στην αγορά, αλλά δεν έχουμε αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό λοιπόν στραφούμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους καλούμε να διεξεγαγούν τις αναλύσεις που έχουμε ήδη ζητήσει. Και την Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά αυτά για να ξέρει τι αποτελέσματα έχει η πολιτική μας. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τωμά θα πάρει τελευταία το λόγο για το 2017 εννοώ. Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει και θα είμαι πολύ σύντομη. Ή, ε, το ελπίζω. Δείχνει ο προπολογισμό αυτός πως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν λειτουργεί. Μπαλώνουμε από εδώ, μπαλώνουμε από εκεί, ε, δεν έχουμε ε, αρκετά κονδύλια, τα παίρνουμε από εδώ να τα δώσουμε από εκεί. Διακόπτει ο κύριος Αρτουή. Ρωτήσατε αν ε, θα ε, λειτουργήσει ως εφαλτήριο ο προπολογισμό το 2017 για την αναθεώρηση του Ποντοπού. Απάντησε το ΜΑ. Ε, μα, έχουμε άλλη μια απόδειξη τώρα. Ήδη από το 2016 είχαμε δει τη διαφορά ανάμεσα αυτά που θέλουμε και αυτά που έχουμε. Από το Brexit θα περάσουμε σε άλλα exit. θα πολλαπλασιαστούν τα exits και μέχρι πού. Δεν λέω ότι είναι το α και το ω των πολιτικών ε, και ότι αυτό σημαίνει ότι είναι ανίσχυρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα, τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω και για το θέμα των πληρωμών αλλά και για το ότι και ίσως να μην έχω καταλάβει, αλλά απευθύνομαι τώρα στους ηγητές ε, Για τον ορίζοντα 2020 και το ΣΕΦ δεν έχουμε αποκαταστήσει τα κονδύλια που περικόπηκαν. Και άρα και κάτι άλλο και πάλι απευθύνω το ερώτημα στου εισηγητές. Δεν έχουμε αποκαταστήσει το ε, τις πιστώσεις ανάλυσης υποχρέωσεων για το Youth Initiative. Και οι υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει δεν ανταποκρίνονται ε, στο, στα κονδύλια του προπολογισμού άβυσος, δεν είναι πλέον διαφορά, χάσμα, ε, διαφορά, άβυσος είναι αυτή που μας χωρίζει από τον προϋπολογισμό και πάμε ε, κατευθείαν να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο, θα πέσει ο τοίχος πάνω μας άμα δεν σταματήσουμε και δεν αναθεωρήσουμε αυτά που κάνουμε. Θα σταματήσω εδώ, ε, Πρόεδρε, όπως λέγατε κι εσείς, Εκπλήσουμε την έλλειψη συνοχή ανάμεσα στι προτεραιότητε ε, του προπολογισμού και τον ίδιο τον προπολογισμό. Μα είμαστε στη χρονιά αναθεώρηση του που και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, αλλά δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Και ε, είπαμε ναι ότι θα είναι το εφαλτήριο για μια ε, ε, προαθεώρηση όχι μόνο του Πουδουπόλα και ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρτουή. Επιτρέψτε μου να επανέλθω ε, στις ε, ε, δυσκολίες που διαπιστώνουμε για την εφαρμογή των υποχρέωσεων των Ταμείων Συνοχής, για το πιλωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση. Βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα το ίδιο δυσκολευόμαστε και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι τόσο περίπλοκη η διαδικασία είναι ε, η πληθώρα των εγγράφων που χρειάζονται, αυτοί που κάνουν αυτά τα πειράματα, είναι τέτοια που περιπλέγει εγώ με τη διαδικασία. Για αυτούς που διστάζουν, ε, μπορώ να πω το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται στις εκλογικές σας περιφέρειες, αλλά εγώ είδα διάφορους ε, φορείς ε, που ε, θέλανε να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια του ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγκαταλείπουν, με τα κύρια ψηλά ακριβώ επειδή είναι περίπλοκες οι διαδικασίες. Είναι σκόπιμο νομίζω να γίνει μια έρευνα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την αυτό το όργιο των διαδικασιών των εγγράφων έλεγχη επιελέγχων από το ελεκτικό συνέδριο. Την κυρία Γκρέσλε, τη φοβερή κυρία γκρέσλ της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Ε, κάποιος πρέπει να ε, βάλει ένα τέρμα σε, αυτή την, ε, σε αυτό το δέδαλο περίπλοκων διαδικασιών. Ξέρω πολύ καλά την κυρία Κρέσλε και συμφωνώ σε πολλά σημεία με την αποτίμησή τη. Δεν πρέπει να κάνει να φοβάται την Επιτροπή Ελεκτών Προπολογισμών και να το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα. Ε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται, γιατί και εμείς δεν συμμετέχουμε 100% στη χρηματοδότηση και πολλοί φορείς δυσκολεύονται να δρομολογήσουν δράσεις διότι πρέπει να δανειστούν για να το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι τροχοπέδι για πολλούς. Ε, συγκεκριμένη έρευνα επιτόπου πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να ξέρουμε γιατί, γιατί δεν ε, προτείνουν προγράμματα οι φορές. Απ' τη μία μας λέει ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν έχουμε επενδύσει. Ε, και τι κάνουμε να φτιάξουμε Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Από την άλλη, εκεί που έχουμε κονδύλια για να γίνουν επενδύσει, δεν προχωράνε τα προγράμματα. Είναι φοβερή η αντίφαση και θα πρέπει να κάνουμε μία έρευνα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη για την παρατήρηση που έκανα. Πρέπει να, γίνουν, καταστούν διαθέσιμα τα κονδύλια που ε, διοχετεύονται κυρίως σε νέου Ευρωπαίου Έρασμου και έρασμου συν. Ε, απευθύνω στους γενικούς συγγητές, ε, απευθύνω αυτή την έκκληση, παρακαλώ, να ε, είναι προσυμφέρον όλοι να προωθήσετε αυτά τα δύο κεφάλαια. Περνάμε στα υπόλοιπα τμήματα. Ο κύριος Ταρά Μα διαφώτισε με, την, ε, με αυτά που μα είπε. Ο ρομπίχ τώρα. Πάολη, θε να μα πει. Τι πιστεύει για το σχέδιο προπολογισμού το 2017, υπόλοιπα τμήματα. Δεν Σας ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι ασχοληθήκαμε πολύ επισταμένως με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ενδιαφέρουσε για μας. Είδαμε ότι τα έσοδα και τα έξοδα στην περίπτωση αυτή διαφέρουν. Υπάρχει απόκληψη. Από πλευρά αρχηγών κυβερνήσεων και κρατών ε, υπάρχει το αίτημα για μείωση των δαπανών και αυτό αναγκαστικά έχει ε, επιπτώσεις και για το προσωπικό και για όλους τους τομείς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και από πλευρά τη ε, επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ποια είναι τα απορίσματα και ποια θα είναι τα συμπεράσματα στα οποία θα πρέπει να βρούμε και εμείς. Merci, Monsieur Ευχαριστούμε, Donado. Ευχαριστώ, ε, η ίδια τάση όπως και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι οικονομίες περικοπές, συρρυκνώνται οι προϋπολογισμοί. Ε, δεν είναι έτσι που θα επιτύχουμε τελικά την πρόοδο στην Ευρώπη και την ανάπτυξη. Έχουμε δυσκολίες πραγματικές για τις πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων και τις πληρωμές κυρίως. Ε, όλοι με τις υποσχέσεις δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στην εφαρμογή έχουμε θέματα. Για τα τμήματα, δύο είναι τα θετικά για μένα. οι μεταφορές ανάμεσα στο το 5 και το 3 για να βγάλουμε 533 εκατομμύρια για την υποδοχή των προσφύγων και ε, τη γραμμή για τα, τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς. Τα υπόλοιπα είναι πιο περίπλοκα. Το είπε ο Ταρά, περιμένουμε διευκρινήσεις πρωτού τοποθετηθούμε κυρίω. Τι γίνεται στην Επιτροπή των Περιφερειών, τι γίνεται στην ΟΚΕ, τι γίνεται στο δικαστήριο, ε, της Ένωσης για το προσωπικό κυρίως. Ε, γιατί κόβουν ε, τις θέσεις, αλλά γίνεται εξωτερική ανάθεση. Άρα δεν έχει κανένα νόημα, λέει ο πρόεδρος. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή θεωρούμε ηλίθιους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, θέλω, θέλω να πάω να τους εξηγήσω. Εγώ πάλι όχι, θα το αποφύγω. Αλλά είναι ιδιαίτερα ανησυχητική ε, η θέση γιατί τι κάνουμε. Είναι μια ανυπόφορη υποκρισία. Τα παίρνουμε από εδώ για να τα δώσουμε από εκεί. μεταφέρω τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί και η εξωτερική, η ε, εξωτερική ανάθεση είναι ότι έχει γίνει τόσο πολύ της μόδας, αναρωτιόμαστε τελικά προ προς τα πού οδεύουμε. Αλλά τα βασικά προβλήματα είναι όπως είπατε και εσείς στο κεφάλαιο, στο τμήμα 3. Ο Σφες δεν ήρθε, ο κύριος Τόρβαλς έπρεπε να φύγει, ο κύριος Σομαχζή δεν μπόρεσε καν να φτάσει. Βάλει δεν είναι εδώ. Δεν έχουμε και... Δεν έχει μείνει και κανένα σκιώδης. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο από σας για τα υπόλοιπα τμήματα. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, η κυρία Καλβίνια, που μας έκανε την τιμή να έρθει, μπορεί να μας διαφωτίσει ίσως. Αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δραστηριότητα τη γραμμή, αν μπορείτε να μας την εξηγήσετε, είναι το μοναδικό περιθώριο λιγμών που έχουν οι ευρωβουλευτές. Ε, Προετοιμάζουν άοκνα, τροπολογίες και εσείς τη συρρυκνώσατε τη γραμμή. Λέγαμε ότι ως επιτοπλίστων θα χρησιμοποιηθεί για την προπαρασκευαστική δράση, για την έρευνα, για την άμυνα. Μήπως τελικά ε, θα περιθωροποιήσετε και θα μας ε, απογοητεύσετε πλήρως ε, με αυτή την πρόταση που κάνετε. Μπορείτε να μας καθησυχάσετε κυρία Καλβίνη. Ευχαριστώ κυρία Αρτουή. Ευχαριστώ όλους τους παριστάμενους. Χαίρομαι για τη σημερινή συζήτηση. Και χαίρομαι για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αναγνώριση των προσπαθειών που κατέβαλε η Κομισιόν. Δεν μας αναγνωρίζεται συχνά η προσπάθεια που καταβάλουμε, γι' αυτό χαίρομαι που επιτέλους ακούω κάτι προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης ε, και αυτό δείχνει ότι συμφωνούμε με τις πολιτικές προτεραιότητες, συμφωνούμε με το πού θα πρέπει να εστιάζει ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Από τις περισσότερες παρεμβάσεις σήμερα βλέπουμε ότι υποστηρίζεται η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Να αναφερθώ στα βασικά θέματα που θέσατε. Να απαντήσω και σε ερωτήσεις σας. Πρώτον, το πρώτο που είπαν πολλοί, το θέμα των πληρωμών. Η πολύ μεγάλη μείωση των πληρωμών. Συμφωνώ κύριε Φερνάντες και με άλλους ομιλητές που λέτε ότι είναι τεράστιο θέμα και λόγος ανησυχίας. Η μείωση των πληρωμών προφανώς οφείλεται σε, στις γενικότερες εξελίξεις που είναι η τελική αρχική φάση της εφαρμογής του παλιού προγράμματος προβλεπόταν ότι είχαμε προβλέψει ήδη στο πολίτες αστυνομικό πλαίσιο το 2017 θα είχαμε μία μείωση, αλλά η μείωση αυτή είναι πολύ πιο υψηλή από αυτή που περιμέναμε λόγω της καθυστέρησης της εκκίνησης των νέων προγραμμάτων. Η καθυστέρηση αυτή έχει να κάνει και με τα διαφορετικά ταμεία, αλλά είναι και στον τομέα της γεωργίας, ίσως γιατί τέθηκε σε ισχύ η νέα ΚΑΠ και καθυστερείται και η εφαρμογή του ΓΕΙ. Πολύ το αναφέρατε. Α, έχουμε μία αργή καθυστέρηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, το ΓΕΙ δηλαδή. Επίσης, ε, θέλετε να σας εξηγήσω και τις καθυστερήσεις και την εφαρμογή. Ε, εμείς υποβάλλουμε εκθέσεις ε, τακτικά και, στις δύο, και στα δύο θεσμικά όργανα για την ε, εφαρμογή και θα καταλάβετε τι γίνεται ε, με την εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2015 και μετά. Τακτικά δίνουμε ε, πληροφορίε στο Κοινοβούλιο και θα το κάνουμε όσον ούπο τι επόμενε μέρε. Σε αυτή την έκθεση θα δείτε το βαθμό τη εφαρμογή, θα δείτε τι καθυστερήσει και επίση θα δείτε ότι δεν περιμένουμε να έχουμε πρόβλημα ε, συσσόρευση δηλαδή ε, καθυστερημένων και απλήρωτων λογαριασμών ε, το 2016. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώ όχι. Φυσικά όπω ε, είπατε πολλοί από εσά, παρά το γεγονό ότι οι πληρωμέ δεν έχουν χαθεί, γιατί έχουμε το συνολικό περιθώριο για τι ε, πληρωμέ, ε, Ευτυχώ έχουμε αυτό το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και επομένω ε, προβλέπουμε κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ανησυχία. Γιατί ε, αργότερα θα, θα μα ζητηθούν να πληρώσουμε αυτά τα ποσά, δηλαδή το 18, 19 και 20. Και επομένως είναι σημαντικό να αποφύγουμε να επαναλάβουμε την κατάσταση όπως αυτή που, προ, που κληρονομήσαμε το 2014. Την περασμένη εβδομάδα θα κάνω την παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού στο Κορεπέρ, εγώ το είπα αυτό τρεις φορές στους ε, πρέσβεις και επομένως μείνετε ησυχοί ότι το Συμβούλιο ξέρει πολύ καλά το κίνδυνο. Αυτή η μείωση που έχουμε στο 2017 να μας στοιχιώσει ε, και να έχουμε περισσότερε αιτήσει για πληρωμέ ε, αργότερα με στο πολιτισμο συνομικό πλαίσιο, δηλαδή το 18-19-20. Περιμένουμε τι προβλέψει τι πληρωμέ ε, τον Ιούλιο από τα κράτη-μέλη και μαζί με την ενδιάμεση αναθεώρηση θα, σας, θα δείτε τι γίνεται για, και τι προβλέψεις έχουμε για το υπόλοιπο πουδουπού. Το φθινόπωρο λοιπόν θα σας δώσουμε μια πιο πλήρη και πιο σαφή εικόνα. Δεύτερο θέμα, ο τίτλος 1. Άκουσα τον τόνο της συζήτησης με ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΥ, που ήταν πολύ πιο θετικό από ότι ένα χρόνο πριν ή έξι μήνες πριν. Ε, ο τόνος αυτός. Από τις παρουσιάσεις που άκουσα εδώ στην Επιτροπή του Προπολογισμού, από τις παρουσιάσεις μάλλον που έγιναν, ε, τελικά ε, καταλάβατε κι εσείς τις θετικές εξελίξεις γύρω από το ΕΦΣΥ. Επίσης ε, υπάρχουν δύο ανησυχίε. Πρώτον η προσθετικότητα και ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια. Ε, αυτό θα το διαμηνήσω τις επόμενες μέρες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το θέμα αυτό της προσθετικότητας. Ε, τώρα, οι προπροσκευαστικέ δράσει για την άμυνα. Συγκεκριμένη ερώτηση. Πώ χρηματοδοτείτε, ο κ. Μαραγάλ το ρώτησε και άλλοι όμω, και πώ ασχολούμαστε με το περιορισμένο περιθώριο που έχουμε στις προπαρασκευαστικές δράσεις. Το ξέρουμε αυτό ότι υπάρχει. Ήταν σκόπιμη η πολιτική απόφαση. Θέλαμε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι έφτασε η ώρα για να βάλουμε επιτάπητος αρκετά λεφτά για να χρηματοδοτήσουμε ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα α, της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί ως πρωτοβουλία της Κομισιόν, ως ένα κλασικό πρόγραμμα για να το πω έτσι, αλλά θα είναι μια χρηματοδότηση ούτω ώστε η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να μπορέσει να συντονίσει τα ερευνητικά προγράμματα τα, και τις προσπάθειες που κάνουν τα 28 κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι είναι και η ώρα να στείλουμε αυτό το σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει αυτόνομη σε ό,τι αφορά την έρευνα στον τομέα της άμυνας και ότι ο στόχος να, βρούμε αυτά τα 25 εκατομμύρια για την προσκευαστική δράση και να τα βάλουμε στο τραπέζι είναι πολύ σημαντικό. Η χρηματοδότηση που προτείνουμε προέρχεται από το α, περιθώριο που έχουμε στο, ε, στο 1α, 15 εκατομμύρια και έχουμε 5 εκατομμύρια από το ΙΤΕΡ και 5 εκατομμύρια από το Κοπέρνικος ε, που θα μπουν στο τελευταίο τμήμα του ΠΟΥΔΟΥΠΟΥ. Δηλαδή αυτά τα ποσά προβλέπονται ε, για την στο Πουδουπού το 2019. Για τον τίτλο 2 έχουν θεθεί ε, κάποιες ερωτήσεις για το περιθώριο ελιγμών που έχουμε. Είναι επαρκής. Τι θα κάνουμε σε περίπτωση κρίσης. Κατά την άποψη Κομισιόν, ναι, είναι επαρκή το περιθώριο του χειρισμού. Γιατί έχουμε 639 εκατομμύρια περιθώριο, που είναι πάνω από επαρκή για να αντιμετωπίσουμε κρίση όπω αυτή που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, μπορέσαμε τελικά να χρηματοδοτήσουμε χωρίς να προσφύγουμε στο αποθυματικό της κρίσης. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ε, αντίστοιχες καταστάσεις όπως η μείωση των τιμών ε, στις παγκόσμιες αγορές, η κρίση του γάλακτος, η απαγόρευση με, με τη Ρωσία κτλ. Αλλά ε, περισσότερο στον τίτλο 5 παρά στον τίτλο 2. Για τον τίτλο 3 τώρα. Ακούστηκαν κάποια σχόλια. Κάποιο μίλησε για την ανάγκη να προχωρήσουμε και στον τίτλο 3. Ε, πού θα ψάξουμε τα λεφτά του τίτλου 3. Θα δείτε στο σχέδιο προπολογισμού πιο πολλέ λεπτομέρειε για την ιδέα χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή ε, συνοριαφυλακή και ακτοφυλακή, ε, το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, την αναθεώρηση του συστήματος στο Δουβλίνο για τους νομίμως ετούντες άσυλο, η νέα υπηρεσία για το άσυλο Υπάρχουν σαφείς στόχοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του στόχου του τίτλου 3. Επίσης, αυτό που είπε ο κ. Ντεπρέ, περισσότερη διαφάνεια για την Ιουλίσα. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω αυτή την απάντηση σήμερα, αλλά θα επανέλθω και θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό της υπηρεσίας Ιουλίσα. Και πολλοί θέσατε ερωτήματα για τις ε, τη νέα, τα νέα κονδύλια, τη μεταφορά ε, μάλλον κονδυλίων για τον τίτλο 4. Αλλά αφού χρησιμοποίησαμε το αποθεματικό για τον τίτλο 3, ε, για τον τίτλο 4 κάπου πρέπει να βρούμε αυτά τα χρήματα. Προσπαθήσαμε να εστιάσουμε, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει και για του πρόσφυγε από την Τουρκία και τιμώντα ε, τι ε, δεσμεύσει απέναντι στο Λίβανο και στην Ιορδανία στην διάσκεψη του Λονδίνου. Το Global Europe είναι ένα τομέα όπου ξέρουμε ότι όσα λεφτά και να είχαμε ποτέ θα αρκούσαν. Αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε ούτω ώστε να βρούμε λεφτά από αλλού με βάση τον οικονομικό προγραμματισμό. Έχουμε και βάλει και μια αναφορά για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες με βάση αυτό που είχαμε σχεδιάσει σε όλο το πουδουπού. Δύο τελευταία λόγια. Για να ευχαριστήσω τον κύριο Αχτουή για την, ε, τον ενθουσιασμό που έχει για την απλούστευση. Και εμένα με ενδιαφέρει τα μάλλον αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί το, και το χρηματοδοτικό κανονισμό και άλλου κανόνε για να το εξασφαλίσουμε. Θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο φιλόδοξοι, ούτω ώστε να υποφελθούμε από την διάμεση έκθεση για να μην διαπραγματευτούμε το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ήδη από τώρα βέβαια, αλλά ήδη σε αυτήν την διάμεσα θεώρηση να σπρώξουμε προ την κατεύθυνση, ούτω ώστε να έχουμε πιο απλό σύστημα για την εφαρμογή του προπολογισμού, που θα μα επιτρέπει τελικά να εστιάσουμε σε αποτελέσματα. Ο κ. Μαραγκάλ είπε ότι είμαστε σε ένα είδος ας πούμε γύρου Γαλλίας, έτσι. Ναι, θα έχουμε βουνά να ανέβουμε μπροστά μας, το βασικό είναι ότι πάντα ο γιος της έχει αίσιο τέλος και ελπίζω και, και εμείς όταν φτάσουμε στη συμφωνία τον Νοέμβριο για το σχέδιο προπολογισμού. Ευχαριστώ. Eh bien, voilà qui est encourageant. Merci. ευχαριστούμε. Είμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γκάιερ. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό το debriefing, σε αυτή την πρώτη ανάλυση για το σχέδιο του 2017, ε, κύριε Τωμά, κύριε Όλμπριχτ, βασιζόμαστε πάνω σας για να διαπιστώσουμε σε ποιο σημείο υπάρχει η σύγκληση και με την αναθεώρηση του Πουδουπού. Και με ένα τέτοιο προπολογισμό θα μπορέσουμε να δείξουμε στους πολίτες, να καταδείξουμε στους πολίτες πόσο απλός είναι ο προϋπολογισμός. Σύντομα ε, θα έχω τη δυνατότητα να σας ε, δείξω ένα έγγραφο για τους προϋπολογισμούς και τους δορυφόρους. Νομίζω ε, ότι όλοι θα ικανοποιηθείτε. Κύριε Γκάι, μήπως θέλετε να αντλήσετε κάποια περάσματα. Ήταν μεγάλη η σημερινή ημέρα. Καλά θα κάνουμε να την κλείσουμε σήμερα. Όλες τις σοφίες μας ε, μπορώ να τις αναφέρω και στην επόμενη συνεδρίαση. Oui, oui. Ça avive le désir. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, la séance est levée.